Okay. Um, welcome everybody. I think we Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Πολύ καλή αυτή η ευκαιρία που έχουμε με, την, με το εργαστήριο μελέτης. Θα σας πω μερικά εισαγωγικά για να αφήσω μετά το λόγο στους ειδικούς που θα μας ενημερώσει, στον Χουάν που θα μας ενημερώσει πρώτα και θα γίνει συζήτηση μετά. Το κέρδος είναι η βάση κάθε εγκλήματος και οι περισσότεροι εγκληματίες προσπαθούν ε, να, παρα... αποκρύψουν τα ε, εισοδήματα, τα χρήματα και τις πηγές της χρηματοδότησής τους. Η νομοποίηση παρανομού χρήματος έχει επιδείξει μεγάλη εφευρετικότητα. Έχει περάσει από τις παραδοσιακές μορφές σε πιο περίπλοκες μορφές νομοποίησης, προσπαθώντας να ξεφύγει από τις αρχές και την προσπάθειά τους να ε, διερευνήσουν και να διώξουν την νομοποίηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Παναμά έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για τέτοιου σκοπούς. Η παρακολούθηση λοιπόν αυτή σε σχέση με, την, ε, με τα έσοδα των εγκληματιών έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι μεγάλη πρόκληση για όλους, δικαστές, εισαγγελείς, επιστήμονες, πανεπιστημιακούς. Αποτελεί νομοποίηση παρανομών εσόδων μεγάλη απειλή για όλο τον κόσμο, αποτελεί απειλή για το κράτος δικαίου, λόγω διαφθοράς ε, δημοσίων λειτουργών και υπονομεύει τις οικονομίες των κρατών. Τεράστιο το κοινωνικό κόστος λοιπόν του εγκλήματος και πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να αναλάβει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτρέψει αυτές τις μεθόδους και τεχνικές που αξιοποιούν οι εγκληματίες. Όταν άρχισα να μελετώ την ε, παρουσίαση που λάβαμε χτες, εντυπωσιάστηκα από τις ε, μεθόδους που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί και ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι με ανησυχεί η κατάσταση όσον αφορά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγεθος των δραστηριοτήτων αυτών και οι πολύ μεγάλες διαφορές και τα κενά δικαίου επίσης στα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε μια μελέτη η οποία έχει πολύ ε, χρόνο και εύρος καλύψει στοιχεία που αφορούν και ε, τις αρχές, διοκτικές, δικαστικές κτλ. και τα συστήματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Εξέτασε η κυρία ε, Ούγκερ. Έχει κάνει μια πολύ εντυπωσιακή δουλειά και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τον καρπό της ε, ανάλυσης και γι' αυτό σας δίνω τώρα το λόγο. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχει να μας πείτε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε που με προσκαλέσατε. Και θα ήθελα σήμερα να σας ε, δείξω τη δουλειά μας και την εντύπωση που έχουμε αποκομίσει από τα από, τις υπερα... από υπεράκτια κέντρα. Η πρώτη φορά που ήρθαμε αντιμετωπίσουμε με αυτό, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η νομοποίηση παράνομων εσόδων. Σας δείχνω εδώ τη διαφάνεια των ΗΕ Εθνών με το πλέγμα που δείχνει έναν ε, λαθρέμπορο ναρκωτικών που συλλέγει το χρήμα από την πόλη των ναρκωτικών, το περνάει στην τράπεζα, μετά από εκεί πάει στις υπεράκτιες τράπεζες και στο τέλος αξιοποιείται το χρήμα αυτό για την αγορά σκαφών, ε, μηχανών, αυτοκινήτων, ακινήτων και άλλων αγαθών για να κρυφτεί. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τέσσερα πράγματα. Καταρχάς ε, τα υπεράκτια κέντρα χρησιμοποιούνται όντως για εγκληματικές, εγκληματικούς σκοπούς. Θα σας ε, δώσω στοιχεία από συνταξιούχο αστυνομικό της Ολλανδίας των κατοχωρών ο οποίος ε, έκανε ένα δακτορικό όταν βγήκε στη σύνταξη μετά θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση της τρίτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων Όπω είπε και ο Πρόεδρο, έχουμε κάνει πολλέ συνεντεύξει, έχουμε συλλέξει πληροφορίε από πολλέ χώρε. Ήθελα να σα δώσω ε, εντυπώσεις, πρώτες εντυπώσεις για την τέταρτη εκδοχή της οδηγίας αυτής που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2017 μόνο στα κράτη-μέλη και τέταρτον θα προσφέρω κάποιες συστάσεις για τον περιορισμό της νομοποίησης παράνομων εσόδων και της φοροαποφυγής με την ευκαιρία των ε, διαρροών των εγγράφων του Παναμά. Καταρχάς τι σημαίνουν αυτά τα υπεράκτια κέντρα δεν ήταν σαφές για μένα τι σημαίνουν. Αν κοιτάξει κανείς την ιστορική πορεία υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, λειτουργίες και ε, απαρχές αυτών των υπεράκτιων κέντρων που ξεκίνησαν το 1920 με τους εγκληματίες του Σικάγο, των Αλκαπόνε και των λοιπόν που προσπαθούσαν από τις Ηνωμένε Πολιτείες όπου ζούσαν να, απο, να βγάλουν χρήματα στο, στο Delaware, το New Jersey και άλλες τέτοιες υπεράκτιες αρχές για να μην ανοιχνεύονται. Στη συνέχεια έχουμε τις υπεράκτιες ε, εταιρείες, τις περιοχές υπό την κατοχή, τη γερμανική, κατοχώρες και Γερμανία. με επιχειρηματικές δραστηριότητες, Ολλανδικές όπως η ε, Unilever και η που προσπαθούσαν εξ αποστάσεως να ε, κάνουν τις ε, επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Ως φοιτήτρια εγώ και μετά την πετρελαϊκή κρίση διαπίστωσα ότι υπάρχουν τα υπεράκτια κέντρα, κέντρα χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής όπως τον Μπαχρέιν. Και ήταν η πρώτη φορά, κάπου στο 1980, άκουσα να γίνεται λόγος για πρώτη φορά, τουλάχιστον στη δική μου προσωπική εμπειρία, ε, για πρώτη φορά ε, να γίνεται λόγος για τα υπεράκτια κέντρα και στη συνέχεια έχουμε τα πραγματικά υπεράκτια κέντρα στη τέταρτη φάση. Τώρα έχουμε δύο αντικρουόμενες απόψεις για το τι συνιστούν οι υπεράκτια κέντρα. Η πρώτη παράθεση λοιπόν που βλέπετε εδώ είναι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια απόκρυψης που εξασφαλίζει σε κάποιον τη δυνατότητα να αποκρύψει την ταυτότητά του, το απόρριτο, με την υπόσχεση χαμηλού φόρου, απορρίτου, μυστικότητας κτλ. Ο άλλος ορισμός λέει όχι, υπεράκτιο κέντρο είναι αυτό το οποίο ε, διεκδικεί την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών, των mutual funds, των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών κτλ. Άρα ένα κέντρο όπως αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα θεωρούνταν ότι είναι υπεράκτιο κέντρο. Άρα πρέπει είτε να επιλέξουμε τον πρώτο ορισμό με παράγοντα ιδιαίτερα το απόρριτο και τη μυστικότητα ή την έννοια της επένδυσης. Και άρα θα τεθεί το ερώτημα αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να θεωρηθεί υπεράκτου κέντρο ή η Φραγκφούρτη. Ή αλλιώς θα βαίνουμε μόνο στον Παναμά και κάποιες νήσους. Εγώ, ναι και δεν γνωρίζουμε περισσότερα, θα προτιμούσα να επιλέξω τον πιο ευρύ δυνατό ορισμό. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τους ορισμούς για το πόσα είναι τα υπεράκτια κέντρα, αναλόγως του ορισμού που επιλέγει κανείς, μπορούμε να έχουμε περισσότερους λιγότερους. Το Δούνο του αρχικά είχε αναφέρει 20 με τον Ρίτσαρτ Μέρφυ που ανέφερε 92 αρχικά, μετά το Δούνο του 69 του 2000. Εγώ θα έλεγα ότι αν περιοριστούμε στα 40 μιας άλλης μελέτης μπορούμε να είμαστε σε κάποια λογικά όρια τα ποσά που διαχειρίζονται και πάλι θα εξαρτηθούν από τον ορισμό και τον εντοπισμό του τι συνιστά υπεράκτιο κέντρο, εάν δηλαδή οι συναλλαγές μέσα στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να συνιστούν ε, υπεράκτια δραστηριότητα. Πάντως έχουμε μεταξύ μεταξύ 3 εκατομμυρίου και 21 τρισεκατομμυρίων σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, με τους δικούς μου υπολογισμούς μπορούμε να πούμε ότι με ασφάλεια ότι έχουμε 7,8 τουλάχιστον 3 εκατομμύρια εδώ είναι ο μακρύς κατάλογος των υπεράκτων κεντρών, 92, πιο μεγάλος, του Ρίτσαρτ Μέρφυ, σε όλο τον κόσμο, πολλές χώρες. Με μπλε και πράσινο αναφέρω, ε, με μπλε και κόκκινο αναφέρω και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά βλέπετε και τον Παναμά και άλλους. Πάντως, ο αρχικός ορισμός με τα υπεράκτια κέντρα είναι πολύ ευρύς από ό,τι βλέπουμε. Τι κάνουν λοιπόν αυτά τα υπεράκτια κέντρα οι επιχειρήσεις. Τι κάνουν. Βοηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητα, στην εξασφάλιση επενδύσεων. Βοηθούν καμιά φορά επιχειρήσεις που για λόγους ανταγωνιστικούς θέλουν να ε, αποκρυφτούν από τους ανταγωνιστές τους και άρα βγαίνουν σε υπεράκτιο κέντρο. Όπως και να έχει το απόρριτο, η μυστικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έστω και για να κρυφτεί κανείς από τον ανταγωνιστή του. Ε, βοηθούν στην φοροαποφυγή. Η απάντηση που θα δώσουμε είναι ναι. Βοηθούν του εγκληματίε και τι οργανωμένε εγκληματικέ ομάδε στο νομοποίηση παρανομών εσόδων και πάλι η απάντηση θα είναι ναι. Ε, μια μελέτη του Ιαν Φαν Koenigfeld, που δυστυχώς είναι μόνο στα Ολλανδικά, πρόκειται για έναν πρώην ε, αξιωματικό συνταξιούχο της ε, ΣΔΟΕ των κάτω χωρών, ο οποίος στη συνέχεια έκανε και ένα διδακτορικό, πάντως έχει δουλέψει στη δίωξη και έχει κάνει πολλές επισκέψεις υπεράκτια κέντρα. Με την ευκαιρία λοιπόν της σύνταξής του ετοίμασε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, διδακτορικό, το, του οποίου τα πορίσματα θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν από αυτό τα μητρώα που εξέτασε ο κύριος Φαν Κόνφελτ όλων αυτών των εταιριών με βάση τις πηγές που δείχνουν 4,2 εκατομμύρια υπεράκτιες εταιρείες. Σε όλες τις χώρες που έχω σημειώσει το χάρτη θα διαπιστώσετε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός υπεράκτων εταιρικών εντοπίζεται στις, ε, στην Αμερικανική Ήπειρο και την Καραϊβική. Στην Ευρώπη έχουμε 687.000, λιγότερα στην Αφρική. Οι όγκοι όμως, οι χρηματικοί που διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Η εκτίμηση, μάλλον θα έλεγα με, απόδειξη, με αποδείξεις ε, εντόπισε ο κ. Φανκόνινφελτ την προέλευση αυτού του πλούτου και τον προορισμό του. Και εδώ βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων από την Ευρώπη, από ευρωπαϊκά κράτη, πάνε σε ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρώπη έχει σε όγκο ε, χρηματικό το μεγαλύτερο ποσό, τα μεγαλύτερα ποσά. Ένα τρισεκατομμύριο στην Ελβετία στη 0,73 εκατομμύρια κάτω χώρε ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Τζέρσεϊ. 3 εκατομμύρια συνολικά από τα 7,83 χρηματικών όγκων που εντόπισε ο κ. Φανικόνφελτ είναι από χώρες της Ευρώπης σε χώρες της Ευρώπης. Άρα δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι δεν μας αφορά το θέμα και ότι αφορά μόνο το τον Παναμά. Οι υπεράκτες εταιρείε έχουν πολύ έντονη δραστηριότητα μέσα στην Ευρώπη, από ευρωπαϊκές χώρες σε ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να εντοπίσω, να εστιάσω την προσοχή σας στην τελευταία στήλη, που βρίσκονται οι ευρωπαϊκές Χώρε, τα ευρωπαϊκά υπεράκτια κέντρα, εκεί που θα πάνε οι Ευρωπαίοι να βάλουν τα χρήματά του. θα δείτε ότι κάθε χώρα έχει τι δικέ τη ε, προτιμήσεις. Οι Γάλλοι Φερρυπίν πάνε στο Μονακό, οι Ιταλοί στο Σαν Μαρίνο, στο Κάμπο Ντιτάλια, οι Ολλανδοί λίγο πιο πέρα την Αρούμπα και τι Ολλανδικέ Αντίλε πρώην απικίε. η Πορτογαλία τη Μαδέιρα, η Ισπανία τη Μελίλα, Μελίλια, το Ρεμάνο Βασίλειο παρουσιάζει εκρηκτικό αριθμό ε, υπεράκτιων κέντρων από τα ε, νησιά της Μάχης, το Guernsey, το Isle of Man, τις Παρθένες νήσους. Πολύ μεγάλο αριθμό λοιπόν και παρότι υποτίθεται ότι είναι πολύ αυστηρή η Βρετανία σε σχέση με τις τραπεζικές ε, ρυθμίσεις δεν έχει μπορέσει να συγκρατήσει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτών στις ε, στα υπεράκτια κέντρα. Άρα τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να στοχεύσει η Ευρώπη, να ξεφορτωθεί αυτή την κατάσταση, να απαλλαγεί από αυτή την κατάσταση. Έχετε και τις λοιπές χώρες νομοποίησης με βάση και έναν δίκτυο. Ε, χρηματοπιστωτικής μυστικότητας. Μια σειρά από χώρες εμφανίζονται στον κατάλογο αυτών. Μπορεί να μην έχει ηγετική θέση σχέση με το ξέπλυμα χρήματος η Ευρώπη, εκτός από το Λουξεμβούργο βέβαια, που έχει μια από τις πιο ψηλές θέσεις, γιατί βεβαίως ε, το Αφγανιστάν και άλλοι εχθροί των ΗΠΑ έχουν ε, θέση πιο ψηλά στον κατάλογο. Αλλά πάντως Ω προ το απόρριτο πάντα, υπάρχουν χώρε που παρουσιάζουν έντονο τέτοιο χαρακτήρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, 28η, χώρες που καλύπτουν με τραπεζικό απόρριτο περισσότερο από ό,τι άλλε αυτέ τι συναλλαγέ. Και άρα γεννούν υποψίε ότι μπορεί να γίνονται και συναλλαγέ ε, των οποίων την προέλευση δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε. Αλλά πάλι θα εστιάσω την προσοχή μου στην τελευταία στήλη με τα νησιά αυτά που έχουν επιλέξει οι ευρωπαϊκέ χώρε για την ανάπτυξη των λιγότερο καθαρών συναλλαγών του. Τι κάνουν λοιπόν αυτά τα υπερακτία κέντρα σε σχέση με του ε, εγκληματίες. Έχει 17 και τις 17 υποθέσεις ε, ναρκωτικών από το 1990 το έως το 2012 ε, αναλύσει ο Φαν Κόνενφελτ με βάση τα στοιχεία του, με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας και του εμπορικού επιμελητηρίου για τις εγκληματικές ε, δραστηριότητες και υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί και διαπιστώνω ότι 741 εγκληματικές υποθέσεις ενέπλεκαν 3.434 334 ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές με όγκο 56 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα τελευταία 14 χρόνια. 56 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για μία χώρα ανοιχνεύτηκαν με τρόπο αποδεδειγμένο για διαχείριση σε υπεράκτια κέντρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για κάτι το ανώδυνο. Πρόκειται για τεράστιου όγκους χρηματικούς και εδώ μιλούμε όχι μόνο για φόρο αποφυγή αλλά για καθαρά εγκληματική δραστηριότητα. Το 80% των δραστηριοτήτων αυτών αφορούν ε, συναλλαγές μεταξύ τραπεζών, άρα έχουν ευθύνη οι τράπεζες γιατί προσφέρουν συμβουλές στους πελάτες τους για τη χρηματοδότηση των υπεράκτιων κέντρων ή που μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους. Άρα είναι απαραίτητο, εάν θέλει κανείς να περιορίσει αυτό το πρόβλημα, να ελεγχθούν οι τράπεζες. Στις κάτω χώρες βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες υπεράκτιων κέντρων ε, που έχουν να κάνουν με την αγορά ακινήτων. Για μικρέ χώρε, βέβαια, η αγορά ακινήτων είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο αγοράζει τα ακίνητα. Όταν πρόκειται για μια υπεράκτια επιχείρηση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο τελικά θα είναι ο κάτοχο αυτού του ακινήτου Ανεπιθύμητη ενδεχομένω, διότι διαφορετικά θα προέβαιναν σε μια νόμιμη αγορά ακινήτου. Και άρα εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Επίση, διαπιστώνουμε ότι από την ε, η εισαγωγή πιο αυστηρών κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εντείνονται οι προσπάθειες που έχουν να κάνουν με τη φοροαποφυγή, τη διαφθορά, τη νομιμοποίηση του χρήματος, τη φοροδιαφυγή μέσω των υπεράκτιων. Δηλαδή, όσο πιο αυστηροί γίνονται οι κανόνες στην Ευρώπη, τόσο εντείνεται η δραστηριότητα προς τις υπεράκτιε εταιρείε. Η Γερμανία, Φερρυπίν, όταν ξαφνικά αναγκάστηκε η Ελβετία να αποκαλύψει στοιχεία ε, τραπεζικών λογαριασμών που διακρατούσε ε, παρουσίασε εκρηκτική ανάπτυξη ο αριθμό των υπεράκτιων επενδύσεων σε άλλα κέντρα που έφευγαν από τη Γερμανία. Μια μελέτη επίση τη γερουσία των ΗΠΑ δείχνει τον αριθμό των ιδιωτών που σχετίζονται με υπεράκτια κέντρα. Και βέβαια και των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων οι οποίε έχουν με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσει την φόρο αποφυγή, περνώντα μέσα από κέντρα από ε, υπεράκτια και οι ιδιώτες βεβαίως ε, μπορούν να χρησιμοποιούν πιο εγκληματικά μέσα. Βέβαια πάντα υπάρχουν όλοι αυτοί οι σύμβουλοι και φοροτεχνικοί κτλ. που τους καθοδηγούν προς τα που θα πρέπει να τοποθετούν τα χρήματά τους. Τι κάνει η Ευρώπη, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα για να αποτρέψει την νομοποίηση παράνομων εσόδων και, τι εγκληματικέ τις εγκληματικές δραστηριότητες. Κάναμε την ανάλυση της τρίτης οδηγίας για την καταπολέμηση παράνομων εσόδων μεταξύ 2009 και 2012. Μια εκτεταμένη έκθεση προέκυψε κατόπιν της αναλύσεως αυτής με ομάδα της Ουτρέχτης. Βλέπετε εμένα αλλά και τέσσερις καθηγητές στα αριστερά ε, καθηγητές του διοικητικού δικαίου από την Αυστραλία, τον Τζον Βόκερ, ποινικολόγο και άλλους. Και εγώ ως ε, οικονομολόγος ήμουν μέλος της ομάδας αυτής. Βλέπετε λοιπόν στα δεξιά τους ε, καθηγητές και στα αριστερά τους φοιτητές μας μια καταπληκτική ομάδα που μας στήριξαν στην ε, προσπάθεια αυτή. Ο ένας μπήκε λίγο αργότερα. Πολλά διδακτορικά προέκυψαν από το project αυτό. Με πολύ ενθουσιασμό λοιπόν δούλεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι επί τρία χρόνια. Είχαμε 200 ερωτήσεις με τις οποίες προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την κατάσταση, μελέτες που αποστήλαμε σε όλες τις χώρες, τις 27, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κροατία, άρα δεν καλύπτεται δυστυχώς από την αξιολόγησή μας. Στείλαμε σε ε, αρχές δίωξης ε, του οικονομικού εγκλήματος, σε υπουργεία, τράπεζες, αρχές εποπτείας της κάθε χώρας, τα ερωτηματολόγια αυτά, τα οποία ε, συμπληρώθηκαν και στη συνέχεια εκπρόσωποι των φορέων αυτών προσεκλήθησαν σε ε, ε, ημερίδες εργασίας με τα Υπουργεία κτλ. για να συζητήσουμε τα πορίσματα και είδαμε αποτελέσματα και για χώρες που δεν θα είχαν ενδεχομένως ενδιαφερθεί αλλά όταν τους ετέθη το ερώτημα είδατε ένα τέτοιο φαινόμενο, διαπιστώσατε με τέτοια συναλλαγή, τότε ναι απάντησαν ε, και διαπιστώθηκαν όλες οι διαφορές με πολύτιμα αποτελέσματα και με πολύ καλή συνεργασία από πλευράς των κρατών. Σε διάφορες ομάδες παρουσιάστηκε αυτό το έργο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να εξασφαλίσουμε και τη συμφωνία των κρατών στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν συνεργάστηκε η Γαλλία. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί την εποχή εκείνη και δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Ιδάλλως όλες οι χώρες που ζητήσαμε συμβολή συνέπραξαν. Πέντε πράγματα θέλησαμε να μελετήσουμε. Καταρχά, αν υπάρχει απειλή από την νομοποίηση παρανομών εσόδων. Άρα, γιατί αν δεν υπάρχει απειλή, δεν χρειάζεται να, να το θεωρήσουμε ω ε, κάτι το επικίνδυνο. Ε, δεύτερον, τι γίνεται σχέση με την υλοποίηση τη τρίτη οδηγία για την νομοποίηση. Τι κάνανε οι χώρε, ε, την αντιγράψαν όπω ήταν στο, ευρωπαϊκό, στο εθνικό του δίκαιο ή το, την προσαρμόσανε. Τρίτον, πώς έγινε η εκτέλεση της οδηγίας, ε, πώς αναπτύχθηκαν ε, οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος, τι έκαναν οι διοκτικές αρχές, οι εισαγγελίες και τι αποτέλεσμα, δηλαδή συγκεκριμένα πόσες καταδίκες προέκυψαν χάρη σε αυτή την ε, νέα οδηγία. Για όλες τις χώρες έγινε η σχετική μελέτη με πρώτο αποτέλεσμα το πόσο ευάλωτες, εκτεθειμένες σε κίνδυνο μπορούν να είναι οι χώρες για το θέμα της νομοποίησης πάντα και βεβαίως υπάρχει και η προβολή σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσματα πάντως σαφέστατα ότι στη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερη η απειλή από ότι στην Ανατολική. Είναι σαφές δηλαδή ότι οι πλούσιες χώρες, αυτές που έχουν ισχυρά χρηματοπιστωτικά κέντρα, μεγάλο ΑΕΠ, εκεί όπου μπορεί να αποκρυβούν, να αποκρυβούν οικονομικές δραστηριότητες και τα χρήματα προκύπτουν από αυτές, πολύ πιο εύκολα είναι πιο εκτεθειμένες στην ομοποίηση παρανόμων εσόδων από αυτές της Ανατολικής Ευρώπης. Παραμένει πάντως, και φανταστείτε τι θα σας πω, σε όλο τον κόσμο πρώτη στη γραμμή η χώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ε, ε, ένα δεύτερο των ποσών που περνούν από νομοποίηση παράνομων εσόδων περνούν μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό και οι αρχές τους ε, έχουν τόσο έντονη δραστηριότητα για την καταπολέμηση της νομοποίησης. Σε σχέση ΑΕΠ τώρα, ως προς το μέγεθος της χώρας, χώρες που έχουν πολύ πιο υψηλό κίνδυνο είναι αυτές της Βαλτικής, με μικρό μέγεθος, ε, και λόγω της ε, ε, εγκύτητάς του στη Ρωσία, όπου είναι εύκολο τα ρούβλια να μετατραπούν σε ευρώ, και βέβαια το Λουξεμβούργο και άλλες χώρες μικρές που μπορεί να έχουν μεγάλες απειλές να αντιμετωπίσουν σχέση με το μέγεθός τους. Στην επόμενη διαφάνεια, οι νομικές Συνέπειε. Η δουλειά που έκαναν οι νομομαθεί μα και κυρίω οι καθηγητέ του διοικητικού δικαίου, το σχεδιασμό τη οδηγία, δηλαδή μελέτησαν και τον τρόπο ε, μεταφορά τη στα εθνικά δίκαια και υλοποίηση τη. Πρώτο, πρώτη ένδειξη. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να περάσει στην εθνική νομοθεσία αυτή η οδηγία. Στι περισσότερε μελέτε λέμε ότι αν έχει περάσει πολλή χρόνο σημαίνει ότι υπήρξε και μεγάλη αντίσταση. Εάν μεταφέρθηκε σχετικά γρήγορα θα ήταν μικρότερη η αντίσταση. Δεν επαληθεύθηκε αυτή η υπόθεση. Ωστόσο σημειώνονται σημαντικέ διαφορέ στη μεταφορά τη οδηγία. Η Γαλλία χρειάστηκε τρία χρόνια. Χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν αμέσω στην ενσωμάτωση τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Όσο πιο μεγάλη είναι η γραμμή ε, η οριζόντια, τόσο πιο πολύ χρόνο χρειάστηκε μια χώρα για να ενσωματώσει το εθνικό δίκαιο την οδηγία. Ρωτήσαμε τους λόγους για την καθυστέρηση αυτή, εκ των οποίων ε, προβάλλονται αρκετές απαντήσεις. Η Ιρλανδία Φερρυπίν μας είπε ότι είχε νομικά εμπόδια να αντιμετωπίσει, γιατί η οδηγία αυτή δεν μπορούσε να εγγραφεί απρόσκοπτα στην ένωμη τάξη της χώρας. Και έπρεπε να βρουν μια λύση για μια οδηγία τέτοια, τέτοιου τύπου. Άλλα προβλήματα ήταν αυτά που κατέγραψαν χώρες όπου αντέδρασαν ε, οι κύκλοι των ε, δικηγόρων, κοινωνική αντίσταση, κάτω χώρες, ε, Ολλανδί, Βέλγιο, Γαλλία και άλλες χώρες αντιμετώπισαν τέτοιου είδου αντιδράσεις. Πολιτικές δυσκολίες επίσης. Το Βέλγιο μας είπε δεν είχαμε κυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της οδικίας. Άλλες δυσκολίες οι μακροχρόνιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη Γαλλία. Αυτό βέβαια δεν μας παρουσιάστηκε σε συζήτηση, αλλά επί χάρτου μόνο. Εκεί πήρε τρία χρόνια η μεταφορά. Ωστόσο, δεν υπήρχε πολιτική αντίσταση από ορισμένε χώρες που είχαν ήδη εισαγάγει τις προδιαγραφές και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν προβλήματα ως προς την εισαγωγή τη οδηγία, γιατί προϋπήρχαν τα συστήματα και εκεί ενσωματώθηκε χωρίς πρόβλημα γιατί είχαν γίνει ενημερώσει ε, τα εργαστήρια συζητήσεων κτλ. Δεν επευλήθη εκ των άνω η νομοθεσία αυτή, αλλά υπήρχε η σχετική προετοιμασία ήδη. Και διαπιστώνουμε ότι τα παλαιότερα κράτη-μέλη έχουν σημαντικά περισσότερε καθυστερήσει από ότι τα νέα κράτη-μέλη. Κάτι που μπορεί να είναι και αισιόδοξο, αλλά και απεσιόδοξο μήνυμα, γιατί διαπιστώσαμε ότι τα νεότερα κράτη-μέλη απλώ έκαναν κοπιπέ τη οδηγίε και έτσι προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα Χωρί αυτό να σημαίνει ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα και το άλλο είναι ότι τα ε, κράτη-μέλη που είχαν εσωτερική εποπτεία με επαγγελματικέ οργανώσεις ε, που αναλαμβάνουν την εποπτεία είχαν καθυστερήσει στατιστικά υψηλότερε, γιατί έπρεπε να περάσουν προσθέσεις διαδικασίε η ενσωμάτωση της οδηγίας. Αυτό λοιπόν χωρί σοβαρές πολιτικές αντιστάσεις όπως είπαμε για την οδηγία και γενικά βλέπουμε ότι υπήρχε μια καλή προετοιμασία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνητικά στοιχεία και αποτελέσματα της οδηγίας. Διαμαρτυρήθηκαν οι χώρες ότι σημειώνονται διαφορές μεταξύ των συστάσεων FATF, για τα, πρότυπα δηλαδή, και της τρίτης οδηγίας. Φερρυπίν, η απλουστευμένη αρχή της πρόληψης και η αξιοπιστία του τρίτου μέρους τα ισόδυναμα Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα λέμε. Εάν δηλαδή υπήρχε μια εσωτερική ε, συναλλαγή από μια χώρα που θεωρούνταν ασφαλής τότε δεν γινόταν επαλήθευση ενώ η οδηγία την απαιτούσε. Άρα μπορεί μια χώρα να τηρούσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά δεν τηρούσε τα ε, πρότυπα FATF. Αντιφάσεις λοιπόν που τους έφεραν ε, δυσκολίες και δυσκολίες είχαν και ως προς την ερμηνεία κάποιων διατάξεων που βέβαια ότι η τέταρτη οδηγία έχει αντιμετωπίσει, έχει λάβει υπόψη, δηλαδή ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης, πώς ορίζεται ο κάτοχος ή ο κύριος, ο δικαιούχος των κονδυλίων. Ε, πολιτικοί που ενδεχομένως ε, εκτίθενται με τα στοιχεία. Στα στοιχεία αυτά έχουμε διαφορετικό χαρακτηρισμό ανάλογα με το αν βρίσκεται ο τελικός αποδέκτης στο εσωτερικό της χώρας ή εκτός αυτής, ή αν είναι politically exposed person, PEP e δηλαδή. Αυτά πάλι τα λαμβάνει υπόψη η τέταρτη οδηγία. Εδώ προτάθηκε, δεν λέω ότι μας ακολούθησαν γιατί υπήρχαν σχετικές προτάσεις και πιο πριν, πάντως άλλαξαν κάποια πράγματα. Ε, δέκα σελίδες από την ε, ανάλυση μας για πολύ μικρά και ασήμαντα θα έλεγα ε, νομικά προβλήματα που μπορεί να έχουν σημασία για τους νομομαθείς αλλά ίσως δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ εσάς και άλλωστε έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και δεν θα είναι πια τόσο ενδιαφέρον. Τα αφήνω λοιπόν τα, τις δέκα αυτές σελίδες της μελέτης και πάω στην επόμενη διαφάνεια που έχει να κάνει με την εκτέλεση. Τι έκαναν δηλαδή οι αρχές δίωξης του εγκλήματος σε σχέση με την οδηγία αυτή. Καταρχάς έπρεπε να συσταθούν αυτές οι αρχές και είχαμε μια μεγάλη ποικιλία ομάδων ε, ε, οικονομικών πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες σε σχέση με οικονομικές συναλλαγές και έπρεπε να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν ε, ε, ε, διοικητικοί υπάλληλοι, ε, υπάρχουν αξιωματούχοι της αστυνομίας με μπλε και ορισμένοι που, είναι, έχουν και τις δύο ιδιότητες και μετά είναι οι δικαστικοί οι οποίοι είναι πιο ουδέτεροι. Δεν είναι τόσο εμπλεγμένοι. Έχουμε λοιπόν ε, διάφορες ε, ε, διαφόρους ενεχόμενους και αυτό το οποίο βρήκαμε είναι ότι είναι πιο σημαντικό ε, πόσο προσωπικό έχουν αυτές οι μονάδες ούτως ώστε να εργαστούν και είδαμε ότι η Γερμανία είχε μόνο 18 άτομα τα οποία να εργάζονται σε αυτή τη μονάδα και αυτό το ποσοστό είναι μικρό, αυτό ήταν εντυπωσιακό και η Ιταλία είχε 100 ανθρώπους, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ήταν τοποθετημένοι στην κεντρική τράπεζα, αλλά δεν είχαν καμία πρόσβαση στην αστυνομία. Ε, τώρα βεβαίως έγιναν κάποιες αλλαγές στην Ιταλία αλλά και στην ε, Γερμανία. Η, ε, από την, υπάρχει μια μετακίνηση από την αστυνομία στη δημόσια διοίκηση, αλλά υπάρχει μια, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον αφορά το προσωπικό και πόσα χρήματα επενδύονται ούτως ώστε για την νομοποίηση των παράνομων εσόδων. Ε, και επίσης ε, υπάρχουν κάποια, κάποιες ειδικέ ε, αρμοδιότητες. Ορισμένοι βοηθούν με το σχέδιο της έκθεσης, άλλοι έχουν εποπτικές δραστηριότητες, άλλοι διατυπώνουν κατευθυντήριες γραμμές, άλλοι διατυπώνουν κυρώσεις, Άρα ε, άλλοι έχουν τεράστιο όγκο εργασία, ενώ ορισμένοι έχουν να υποβάλουν κάποιε εκθέσει, να διατυπώσουν κάποιε εκθέσει και να τι ε, διαβιβάσουν στην αστυνομία κλπ. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ε, διαφορετικά προφίλ απασχόλησης μέσα στις μονάδες αυτές και μπορούμε να δούμε τη διάχυση αυτών των δραστηριοτήτων. ανατολικά είναι πολύ πιο ειδικευμένες, περισσότερες δραστηριότητες από ό,τι δυτικά και είναι πιο σημαντικό να δούμε ε, ποια είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες. Εάν ε, θέλω να βρω ποιος κάνει το ξέπλυμα των χρημάτων, πρέπει να έχω πληροφορίες από την αστυνομία, από τις φορολογικές αρχές, από εμπορικούς ε, φορείς, από την αγορά κινήτων κλπ. κλπ. Εάν υπάρχει κινητικότητα των εγκληματιών σε όλους τους τομείς και εγώ ως μονάδα ε, Τη οικονομική υπηρεσία για τις μυστικέ πληροφορίε που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να συγκεντρώσω μια πληθώρα στοιχείων. Και υπάρχει και το βελικό μοντέλο όπου κατά βάση έχουμε ένα αξιωματούχο σύνδεση, το οποίο δείχνει ότι η βελική μονάδα έχει πρόσβαση στην αστυνομία άρα ε, υπάρχει μια άμεση διασύνδεση με την αστυνομία αλλά εάν ε, δεν έχει κανείς ε, ειδικέ πληροφορίες όπως είναι ε, τα στοιχεία σχέση με τη φορολογία γιατί σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στα, στα, στις φορολογικές δηλώσεις, στα στοιχεία της εφορίας γιατί υπήρχαν χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, δεν υπάρχει τέτοιου είδου πρόσβαση σε αυτά τα φορολογικά στοιχεία. Άρα δεν ε, μπορούμε να έχουμε τέτοια στοιχεία σε σχέση με την νομοποίηση των παράνομων εσόδων, γιατί και εκείνη την εποχή η φοροαποφυγή δεν συνδεόταν με το ξέπλυμα χρημάτων. Αλλά αυτές οι μονάδες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη βάση δεδομένων εάν θα πρέπει να ελέγξουν διεξοδικά αυτούς που ασκούν την νομοποίηση των παράνομων εσόδων. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η υποπτία. Προσπαθήσαμε να δούμε πόσο, ε, πώς εποπτεύεται η υποβολή αναφορών για τις τράπεζες, για τις υπηρεσίες ε, επιχειρήσεις ακινήτων κλπ. Και εδώ υπάρχουν επίσης διάφορες ε, μορφές εποπτείας στις διάφορες χώρες. Σε ορισμένες είναι ακριβώς ε, αυτή η μονάδα η οποία είναι υπεύθυνη. Σε άλλες χώρες είναι οι νομικές ε, αρχές. Ε, υπάρχει διάκριση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών ιδρυμάτων. ναι, ε, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία στην... Ε, υπάρχουν ποικίλε μορφές μάλλον εποπτείας. Και ε, η πόνοιά μα ότι δεχομένω θα είχαν αλλάξει τα πράγματα δεν επαληθεύτηκε. Για παράδειγμα, οι τράπεζε, οι των τραπεζών δεν μπορούσαν να ανοιχνεύσουν το ξέπλυμα χρημάτων Η εποπτεία είναι κάτι το οποίο λοιπόν θα πρέπει να ε, ενισχυθεί ε, καθώς και η επιβολή κυρώσεων και προστήμων. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή, τι κάνει η αστυνομία και η Γενική Εισαγγελία ειδικότερα. Έχουμε δύο συστήματα στην Ευρώπη. Έχουμε μια ε, νομολογία του αγγλοσαξονικού δικαίου στη Μάλτα και βλέπουμε εδώ ότι ο ρόλος της Γενικής Εισαγγελίας είναι διαφορετικός. Εδώ διεξάγονται μόνο οι ανακρίσεις πριν γίνει η προσαγωγή στο δικαστήριο. Γιατί έστω και αν ένα εγγελέας έχει πάρα πολλέ ε, υποθέσει και ο δικαστή ε, δεν είναι αρμόδιο για τέτοιου είδου υποθέσει για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, ε, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Στο public law υπάρχει μια, γίνεται μια προανακριτική έρευνα Υπάρχουν, λοιπόν, υπάρχουν αυτά δύο διαφορετικά συστήματα τα οποία ισχύουν στις χώρες. Αλλά η Γενική Εισαγγελία στο αγγλοσαξονικό δίκαιο έχει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει. Τώρα, υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων. Ε, όσον αφορά την ποινή φυλάκισης και τα, προ... και τα... και τα χρήματα πρέπει να πληρώσει κανείς. Ορισμένες χώρες έχουν ισόβιες ποινές, ε, άλλες έχουν ε, πέντε χρόνια, προβλέπουν φυλάκιση. Υπάρχουν λοιπόν τεράστια διαφορές μεταξύ των χωρών. Το ποινικό δίκαιο προβλέπει διάφορες ε, Ποινέ για την χρηματοδότηση τρομοκρατικών πράξεων και για την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Εάν δούμε πόσοι άνθρωποι έχουν ε, καταδικαστεί και εδώ έχουμε πράγματι εντυπωσιακά αποτελέσματα και απογοητευτικά θα έλεγα. Όλες αυτές οι προσπάθειες ε, που είδαμε, ε, τις υποβολές αναφορών, την Γενική Ασυγγελία και την αστυνομία κλπ όλες αυτές οι προσπάθειες τελικά όλη αυτή η αλυσίδα προσπαθειών κατέληξε σε εξαιρετικά ισχνά αποτελέσματα όσον αφορά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Η μόνη χώρα η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα είναι η Δανία. Αλλά οι Δανείοι λένε ότι τους υποβοηθάει πάρα πολύ το, ο νόμος τους ε, μπορούν ε, να ασκήσουν ποινικέ ε, διώξεις πολύ πιο εύκολα ενώ στα άλλα νομικά συστήματα πρέπει να αποδειχθεί ότι κάποιος έχει διαπράξει το έγκλημα. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Ενώ στη Δανία κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Ε, γι' αυτό ε, σε ορισμένες ε, χώρες η δίωξη αυτών των εγκλημάτων είναι κόλαση, ενώ για άλλες είναι πραγματικά πολύ εύκολη. Ε, ε τώρα όσον αφορά την αντιστροφή του βάρους απόδειξης υπάρχουν νομικά συστήματα όπου πρέπει να ε, γίνει αυτή η αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Δηλαδή, ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει εκείνος ότι είναι αθώος και όχι ο δικαστής ότι είναι εγκληματίας. Ε, οι καταδίκες ε, πάντως εν γέννη είναι πολύ λίγες Στη Γερμανία έχουν πολύ, ε, όπως σας είπα, περιορισμένο προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Εάν κανείς ήθελε να κάνει αυτή την εγκληματική πράξη, πού θα πήγαινε στην Ευρώπη. Προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες μετρήσεις, κάποιου υπολογισμού και είδαμε. Αυτή είναι η σύσταση προς τους, αυτούς που θέλουν να κάνουν ξέπλυμα χρημάτων. Αυτές τις χώρες που βλέπουμε εδώ με φούξια. Στη, στη Δανία έχουμε πολύ αποτελεσματική διαδικασία δίωξης, αλλά πολύ χαμηλά πρόστιμα So clearly Στη Ρουμανία ισχύει το ακριβώς ε, αντίστροφο. Ωραία λοιπόν. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, πώς μπορεί να δουλέψει η διεθνή συνεργασία μεταξύ, σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητε. Δεν εξετάσαμε το πώς λειτουργούν τα υπουργεία, αλλά οι FIUs και οι γενικές εισαγγελίες των χωρών. Δεν υπάρχει επικοινωνία, για παράδειγμα, μεταξύ των μονάδων αυτών και της Γενικής σας Εισαγγελίας, γιατί υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας των δεδομένων και λοιπά απορρίτου. Εάν η Europol, η Interpol, ε, ε, βεβαίως μπορεί να έχει μία ανταλλαγή στοιχείων με, τις, ε, με την FIU και η, γενική και οι εισαγγελείς επίσης μπορούν να προβούν σε μια ανταλλαγή στοιχείων. Ε, Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι αυτές οι μονάδες μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές και όσον αφορά τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας. Ποια είναι όμως τα εμπόδια ε, στη συνεργασία αυτή όσον αφορά τα αποτελέσματα. Οι περισσότερες χώρες και αυτό το είδαμε στα εργαστήρια. 15 χώρες μέλη έχουν πολλές χρονικές καθυστερήσεις. Όταν ζητήσω μία πληροφορία για κάποιο ύποπτο, αυτό θα έχει εξαφανιστεί πριν πάρω εγώ την πληροφορία. Και πολύ συχνά ε, νομικά κείμενα χρειάζεται πρώτα να μεταφραστούν. Ε, και οι εισαγγελείς ε, θέλουν να έχουν πολύ ακριβή, με ακρίβεια διατυπωμένα κείμενα για την εργασία τους και αυτό είναι χρονοβόρο. Ή πολλές ε, χώρες όπως Οι Ελβετία σου απαντούν ήδη την επομένη με μεγάλη ευγένεια αλλά δεν είναι η απάντηση που θέλαμε ή από την αρχή που θέλαμε. Ε, πολύ συχνά λοιπόν δεν ε, παρέχεται αυτό το οποίο ζητείτε. Και ή πολύ συχνά η προστασία δεδομένων είναι ένα λόγο για τον οποίο δεν δίδεται ακριβή απάντηση από την άλλη χώρα και αυτό συνιστά εμπόδιο. Και η γλωσσική φραγμή σε ορισμένε χώρε είναι ένα εμπόδιο, δηλαδή αν κανεί δεν ομιλεί τη γλώσσα τη άλλη χώρα και πρόκειται όπως είπαμε για νομικά κείμενα τα οποία θα πρέπει να είναι συντεταγμένα σε μια ακριβή γλώσσα και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Μας ε, ε, εξέπληξε όταν ε, καλέσαμε τις χώρες να μας πούν κατά πόσο μια δραστηριότητα συνιστά ξέπλυμα χρημάτων ή όχι. Για παράδειγμα, έχουμε έναν ληστή ε, τα χρήματα τα οποία έχει είναι αυτοξέπλημα. Η Ολλανδία θα πει ναι. Επίσης υπάρχει μιες, ε, υπάρχουν μέσα χώρες οι οποίες κάνουν οι ίδιες όπου ο εγκληματίας κάνει ο ίδιος την νομοποίηση των παράνομων εσόδων. όλες αυτές οι χώρες ε, πρέπει να, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν την νομοθεσία τους. Το self-laundering. Self-laundering can also be uh, convicted. So these things... Η αυτονομιμοποίηση των παράνομων εσόδων λοιπόν θα θεωρηθεί μελλοντικά παράνομη. Ε, τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας, εδώ η εικόνα είναι πιο ομοιογενής. Και εδώ οι ορισμοί είναι πιο ξεκάθαροι. Και μόνη διαφορά είναι κατά πόσο οι προθέσεις επίσης είναι καθοριστικές ή όχι, κατά πόσο γνωρίζει κανείς ε, πού πάνε τα χρήματα κλπ. Αλλά υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση εναρμόνισης ή σύγκλησης ως προς το τι θεωρείται νομοποίηση παράνομων εσόδων και τι όχι. Τέλος, αξιολόγηση πόσο ε, καλή είναι αυτή η πολιτική και πόσο εφαρμόζεται. Αξιολογήσαμε τις χώρες βάσει όλων των κριτηρίων που είχαμε στο project αυτό και αν μια χώρα έχει μόνο ε, πράσινο, τότε είναι τέλεια. Και η μόνη η οποία είναι εντελώς ε, πράσινη και η οποία δεν χρειάζεται να βελτιώσει τίποτα βάσει εξολόγησή μα είναι η Δανία. Όλε οι άλλε χρήζουν βελτιώσεων. το Ηνωμένο Βασίλειο, την ε, πληροφόρηση, την ε, ενημέρωση μεταξύ FIU και γενική εισαγγελία. Άλλες χώρε θα ε, μπορούσαν να κάνουν άλλες βελτιώσεις. Τελευταίο σημείο εδώ στη διαφάνεια, στη στήλη μα, ο αριθμός των καταδικών. Ε, η κάθε χώρα μπορεί να φέρει κάποιες βελτιώσεις. Θεωρήσαμε ότι είναι πιο σημαντικό να καταδείξουμε σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να γίνουν οι βελτιώσεις για την κάθε χώρα. Τώρα, εάν πάρουμε όλα όσα κάναμε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, και τα βάλουμε σε έναν υπολογιστή και θέλουμε να κάνουμε μια cluster ανάλυση και να πούμε ποιε είναι οι ομοιότητες μεταξύ των χωρών και κάνουμε τέσσερι ε, κατηγορίε. τότε το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε τέσσερι ομάδε εντό τη Ευρώπη για την ομοποίηση παράνομων εσόδων. πρώτες είναι, ε, η πρώτη ομάδα είναι αυτές που κάνουν αυτονομιμοποίηση παράνομων ε, εσόδων. Ε, υπάρχει ένας κατάλογος της FATF που αποκλεί τις συναλλαγές με την Αμερική. Το, η δεύτερη ομάδα ε, είναι η ομάδα χωρών που έχουν περισσότερα εσωτερικά προβλήματα, το Βέλγιο, η Ιταλία, χώρες που υφίστανται μεγάλες εσωτερικές, μεγάλες εσωτερικές πιέσεις και όπου η νομοποίηση με εισόδων δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που έχουν οικονομικά προβλήματα κλπ. Η, άλλη ομάδα είναι οι ομάδες που κατακλείζονται όπως η Κύπρος, το, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο που κατακλείζονται από ροές ε, χρημάτων που προέρχονται από παράνομες ε, πηγές και θέλουν να τα νομιμοποιήσουν. Και η τέταρτη ομάδα είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ορισμένες χώρες ήταν εντελώς καινούριο αυτό το φαινόμενο. Χρειάστηκε να συστήσουν ένα νέο τραπεζικό σύστημα και να κάνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και σε πολλά άλλα πράγματα όπου η δραστηριότητα αυτή της νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, δεν ήταν ε, η προτεραιότητά τους. Και πολλές από αυτές δεν ήταν από τεχνική άποψη σε θέση να σχεδιάσουν μια δική τους νομοθεσία για την νομοποίηση των παράνομων εσόδων. Και δεν είχαν και την εμπειρογνωμοσύνη. Ούτε και την απαραίτητη ε, νομοθεσία. Ε, σε, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας μου είχε πει ε, κάποια στιγμή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ε, τους ε, ε, νόμους οι οποίοι θα βοηθούσαν στην καταπολέμηση ομοποίησης παρανόμων εισόδων. Επίσης μου είχε πει ο ίδιος Εισαγγελέας ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν το ρυθμό των άλλων χωρών, των χωρών της Δυτικής Ευρώπης που επί πολλά χρόνια ε, είχαν σκύψει πάνω στο θέμα αυτό. Επομένως, τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες ε, υπάρχουν και θα είναι δύσκολο να υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική. Επίσης, ε, εάν κανείς καταλήξει σε μία και μοναδική προσέγγιση, τότε θα είναι γραμμένη στα βιβλία, αλλά δεν θα ισχύει στην πραγματικότητα. Η τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του, της παράνομης νομιμοποίησης, της νομιμοσύνης <laughs> ποιήσης παρανόμων εισόδων, είναι περίπου ίδια με τις προηγούμενες. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο με προβληματίζει λίγο αφορά την φοροδιαφυγή γιατί αναφέρεται σε tax crime ε, το οποίο θα πρέπει να ονομάζεται πλέον ε, κανονικό ε, έγκλημα. Εγώ δεν είμαι ποινικολόγος ναι, αλλά αναρωτιέμαι ε, τι σημαίνει αυτό σε χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικό νομικό σύστημα, σαν αυτές δηλαδή που ανέφερα προηγουμένως. Ε, κοιτάξτε, εάν η φόρο αποφυγή είναι απάτη, ε, εάν αυτό θεωρείται απάτη, τότε έτσι θα έπρεπε να αναφέρεται και στην τέταρτη οδηγία. Η, η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε κάποια πραγματική αλλαγή. Για την Αυστρία, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οποιοδήποτε έχει αποφύγει, έχει φόρο διαφύγει για πάνω από 100.000 ευρώ, ε, τότε θα έχει υποπέσει σε απάτη και επομένως ε, ε, απάτη, άρα δεν αλλάζει και τίποτα για την Γερμανία που είναι αυτή η οποία ανακοίνησε όλη αυτή την διαδικασία εάν έχει κανείς ε, φόρο ε, αποφυγή για πάνω από 500.000 ευρώ θα μπορούσε να πάει ας πούμε στην Γερμανία. Ε, για τους, για τους Γερμανούς μπορεί Μπορεί να θεωρηθεί πλέον η φοροδιαφυγή ε, για τέτοια ποσά ε, σοβαρό ε, αδίκημα και επομένως ενδεχομένως για τους Γερμανούς να κάνει κάποια διαφορά και σε αυτή την περίπτωση στη Γερμανία μπορεί να υπάρξει ποινική διαδικασία. Επίσης, ε, ενώ στην Αμερική υπάρχει μια κοινή ορολογία στην ε, Ευρώπη ε, πραγματικά τα πράγματα είναι διαφορετικά και επομένως θα πρέπει κανείς να δει στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι ακριβώς σημαίνει tax crime, τι περιλαμβάνει ο όρος tax crime και μια αποσαφήνιση νομίζω ότι θα βοηθούσε έτσι ώστε να κλείσουν κάποια κενά. Έχουμε ε, αυτή τη στιγμή πολλά ε, ε, στοιχεία νομοθεσίας. Έχουμε όπως προερχόμαστε και από μια κατάσταση όπου όπως σας είπα και προηγουμένως έχουμε πολλά νομοθετήματα τα οποία ασχολούνται με το θέμα. Για μία ακόμα φορά το import έρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Αμερικανοί ήθελαν ε, να καταγράφονται και να είναι διάφανες μέσω της ε, σχετικής νομοθεσίας ή ε, διαδικασίες. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα συζητούμε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και ένα σωρό άλλα πράγματα έτσι ώστε να γίνει όλο και λιγότερο δυνατή η φοροαποφυγή στις χώρες. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα αποτελέσματα τα πάντως βλέπουμε ότι επιταχύνονται οι ε, κανονισμοί, επιταχύνεται ε, το νομικό πλαίσιο, πάει όλο και πιο γρήγορα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και ένα project για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έτσι ώστε μαζί με τον Ρίτσαρτ Μέρφυ ας πούμε, και το, τη σχολή της Κοπενχάγης να προσπαθήσουμε ε, να δούμε τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι νέες ε, ε, διεθνείς οδηγίες ή κανονισμοί σε, σε όλες τις χώρες. Να δούμε δηλαδή ποιες τρύπες ας πούμε θα κλείσουν και ποιες άλλες, ποια άλλα κενά θα ανοίξουν. Γιατί στην ουσία αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να ταυτοποιούνται όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα κενά, ε, τα οποία, τα holes τα οποία επιτρέπουν ε, ε, την αποφυγή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ε, ποιες θα είναι οι νέες στρατηγικές τις οποίες ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να βρουν ε, οι ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης ε, οι υψηλού προφίλ εγκληματίες προφανώς θα προσπαθήσουν να βρουν νέους τρόπους. λίγο ακόμα και τελειώσαμε. Έχω φτάσει στα συμπεράσματα. Ε, πρέπει να υπάρξει πραγματική συμμόρφωση όσον αφορά ε, την ε, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Δηλαδή μεταξύ των χωρών, μεταξύ των Υπουργείων, μεταξύ των Γενικών Εισαγγελέων, των δικαστηρίων, σε διεθνές επίπεδο χρειάζεται πολλή συνεργασία και σε μεγάλο βαθμό γιατί τα συμφέροντα είναι κοινά δεν ε, ε, ε, εδώ εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει θύματα ή μάλλον καλύτερα δεν έχει άμεσα θύματα. Οι δημόσιοι κατηγοροί μας λένε συχνά, οι γενικοί εισαγγελές μας λένε συχνά ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στα δικαστήρια σε πολλές φορές με τέτοιες περιπτώσεις γιατί δεν υπάρχει άμεση ε, επίπτωση στο δημόσιο χρήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ξέπλυμα αυτό ε, να γίνει ε, στρατηγικός στόχος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει οπωσδήποτε ζημία, αλλά η ζημία δεν αποδεικνύεται και εν πάση περιπτώσει δεν αποδεικνύεται ως έχουσα άμεση ε, ε, σχέση με την ε, ε, ένα πράγμα είναι ε, το να αντιμετωπίσει κανείς και να καταπολεμήσει ας πούμε το λαθρεμπόριο ή ε, το οργανωμένο έγκλημα ή οτιδήποτε και άλλο πράγμα είναι το θέμα του ξεπλήματος παρανόμων εσόδων κτλ. αυτό που θέλουμε, θέλαμε σε αυτή την έρευνα, στα πλαίσια της οποίας αναλύσαμε οποιαδήποτε συναλλαγή μας φαινόταν ύποπτη, οποιασδήποτε αναφορές συναλλαγών ύποπτες κτλ. Αυτό που θέλαμε είναι ε, να υπάρχει ειλικρίνεια, ε, να μην, ε, να μην κανείς λέει ψέματα σε αυτές τις περιπτώσεις εάν πραγματικά θέλετε ε, να μην ε, αν θέλετε να, να αλλάξει κάτι, δεν αρκούν ε, οι στατιστικές ή τα reports ή οι αναφορές που θα κάνουν οι τράπεζες. Οι αριθμοί, είτε είναι υψηλοί είτε είναι χαμηλοί, δεν μας λένε πάρα πολλά πράγματα. Ε, κάποιες εκθέσεις μπορεί να μας λένε ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ε, καταπολέμησης ε, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν, δεν γίνεται σωστή δουλειά. Δηλαδή δεν πρέπει αυτές οι αναφορές να εκλαμβάνονται ως κριτήρια αξιολόγησης. Εμείς, εμείς μελετήσαμε και αναλύσαμε προσεκτικά όλες τις αναφορές. Έχω και ένα τελευταίο ε, το οποίο, μια τελευταία διαφάνεια που αναφέρεται σε τέσσερις διαφορετικές ε, ομάδες χωρών. Όπως έλεγα και προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν ένα μοντέλο να ισχύσει για όλους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η καταπολέμηση της, ε, του, της ομοποίησης των παρανόμων εσόδων δεν είναι γέννημα ευρωπαϊκό. Έχει έρθει από την άλλη πλευρά του ωκεανού και πολλοί αναφέρονται από τη δική, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σαν ε, ε, τον ευρωπαϊκό τρόπο, την ευρωπαϊκή ανταπόκριση ας πούμε στο ίδιο πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο ε, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη ακριβώ την πολυμορφία τη ε, της Ευρωπαϊκής ε, την πολυμορφία των νομικών συστημάτων, των θεσμικών συστημάτων, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικές πολιτικές αλλά ο στόχος να είναι ίδιος και κοινός. Το πιο σημαντικό είναι να βρούμε ένα σύστημα μεγαλύτερης διαφάνειας ε, και ε, διαφανών συναλλαγών μεταξύ των, και στοιχείων μεταξύ των χωρών μιλών. Νομίζω ότι από πλευράς κανονισμών και ρυθμίσεων έχουμε αρκετά. Ε, το θέμα είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, διεθνή συνεργασία, πρόσβαση σε Μητρώα, γνώση των πραγματικών κατόχων κλπ. Επίσης το να κατονομάζουμε και να κατηγορούμε, ε, να κατονομάζουμε ε, τους υπευθύνους name and shame δεν είναι και η καλύτερη ε, διαδικασία. Το θέμα είναι να ξέρει κανείς πληροφορίες από άλλες χώρες, αυτόματα να... Δηλαδή δεν με ενδιαφέρουν ε, όλα τα ονόματα, με ενδιαφέρει ένα όνομα το οποίο ε, μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικά κομπιούτερ και σε διαφορετικές, ε, σε διαφορετικές λίστες. Αντα, ε, ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμέν, με συγκεκριμένο τρόπο ε, και μεγάλη διαφάνεια. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά ε, νομίζω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ, καλό στοιχείο. ξέρουμε ότι οι εγκληματίες μια χαρά συνεννοούνται μεταξύ τους και επικοινωνούν, άρα και εμείς από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχουμε μια αντίστοιχη ικανότητα διαφανούς και αποτελεσματικού Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Ουγγέρ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση της μελέτης σας και των συστάσεων. Θα ακούσουμε τώρα βουλευτές πρώτα απ' όλα, αλλά και επειδή δεν είναι πολλοί βουλευτές και άλλους παρεμπισκομένους. Ε, Γιάννα Γκόμες. Ευχαριστώ όντως τον συναρπαστική παρουσίαση. Θα χρειαστεί να τη μελετήσω πολύ προσεκτικά γιατί βλέπω να αντιστοιχεί σε πολλές από τις προσωπικές μου παρατηρήσεις από την ίδια μου την πατρίδα, την Πορτογαλία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η νομοθεσία, οι ρυθμίσεις, αλλά η τήρηση, η εφαρμογή τους. Και αυτό βέβαια εξαρτάται και από τους πόρους, ανθρώπινους και τεχνολογικούς, όχι μόνο σε σχέση με τις ε, αρχές ε, που είναι υπόχρεες για ενημέρωση της FIU, αλλά και τις λοιπές ε, που, που έχουν την διερεύνηση οικονομικών πληροφοριών, μυστικών πληροφοριών, αλλά και γενικά τις αρχές. Επί παραδείγματι, στη χώρα μου, είναι ξεκάθαρο ότι η πιο γνωστή ΠΕΠ της Αγγόλας, κυρία Βάλτερ Σάντος, που είναι η κόρη του Προέδρου, δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό στην κάτω, στις κάτω χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Αλλά στην Πορτογαλία μπορεί να αγοράσει τράπεζα, μπορεί να έχει δική της τράπεζα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο και πολύ μεγαλύτερο και σε επίπεδο εποπτείας που δεν φέρνει αποτέλεσμα και σε επίπεδο συνομόρφωσης. Και μιλάμε για πολύ απλά πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση και Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική η δίωξη της νομοποίησης ξεκινώντας από το βασικό έγκλημα, το predicate ε, offense, αλλά και γενικότερα πρέπει να μην επιτρέπουμε στο οργανωμένο έγκλημα συμπεριλαμβανομένης και της τρομοκρατίας να νομοποιεί τα έσοδά του. Αυτό πρέπει να τονίζουμε όλο και περισσότερο, γιατί οι κυβερνήσει μα, δηλαδή, είναι τέτοια η χαλαρότητα προ την εφαρμογή τη νομοθεσία στη χώρα μου, που μπορώ να την αποδώσω μόνο στην απόλυτη αδιαφορία μέχρι συνενοχή των αρχών που ε, έκλειναν τα μάτια. Και δεν μιλώ για τι αρχέ τη Πορτογαλία, μιλώ για τι ευρωπαϊκέ αρχέ. Πρόσφατα που ήμουν στη Μαδέρα, να ενημερωθώ για, τις για την ε, υπεράκτεια εκεί, που δεν θέλουν βέβαια να ακούνε τη λέξη υπεράκτεια, στη Μαδέρα προφανώς. Γιατί η αρχική άδεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγκαθίδρυση το 86-87, αυτού του διεθνού Κέντρου Επιχειρήσεων όπως το ονομάζουν, ε, ρητά λέει ότι δεν τους επιτρέπει να ε, συστήσουν υπεράκτεια. Αλλά μπορούν να κάνουν ό,τι εν γέννη πράττει μια υπεράκτια επιχείρηση. Ο Πίτερ Σάδερλαντ, ο Μπαρόζο, που αμέσως μετά βέβαια πέρασε στην ε, Goldman Sachs και μάλλον είναι ο μεγάλος ειδικός της νομοποίησης, ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη σχετική άδεια και άρα επέτρεψαν κάθε τέτοια δραστηριότητα υπεράκτειας. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν κοιτάξουμε τις ε, αμνηστεύσεις τις φορολογικές που δόθηκαν στη χώρα μου, ιδιαίτερα μετά την κρίση 2005, 10, 12, τρεις διαδοχικές φάσεις, εδώ πρόκειται ακριβώς για νομοποίηση μέσω της νομοθεσίας των παράνομων εσόδων. Το 12. Αυτοί που είχαν χρήματα στην Ελβετία, στα Καϊμάν, με 7,5% μόνο φόρο, ξεπλένονταν από κάθε αδίκημα ενοχή και, όχι, και ούτε καν χρειάζονται να ξαναφέρουν τα χρήματα στην χώρα. Και αυτά κάτω από τη μύτη της λεγόμενης Τρόικα. Ή τέλος πάντων αυτών των αρμόδιων για την προσαρμογή, όπως λέγεται. Πιο σωστά. Δημοσιονομική προσαρμογή. Τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της παρανομής. Εσείς πιο πολύ μιλήσετε για την τρίτη, αλλά στην τέταρτη ο Επίτροπος μας είπε ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η ρήτρα στην πρώτη οδηγία, ότι αν τυχόν δεν μπορέσει να ανοιχνευθεί ο κάτοχος, τότε θα πρέπει να καταγράφει τουλάχιστον ο κυριστής. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, αν είναι σύσταση του ΦΑΤΦ, τον ΦΑΤΦ ή όχι. Είναι λάθος αυτό γιατί αφήνει παραθυράκια. Το πρώτο πράγμα που πέρασε από την οδηγία, την πρώτη οδηγία, στην εθνική νομοθεσία στην Πορτογαλία από την προηγούμενη βέβαια κυβέρνηση, ήταν ακριβώ αυτό το άρθρο, αυτή η ρήτρα. Γιατί ήταν αυτή που άνοιγε τα παραθυράκια και επέτρεπε την νομοποίηση, όπω βέβαια την εννοούσε και η Τρόικα, και έτσι μπορούσε να αποκρυφτεί ο ε, κάτοχο και δικαιούχο. Και θα ήθελα να συστήσουμε κάτι το οποίο όλοι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρνηθεί για χρόνια να κοιτάξουν τις λεγόμενες χρυσές βίζες και προγράμματα επενδύσεων. Δεν είναι αυτό ένα μέσο ενεργού ξεπλήματος παράνομων εσόδων, νομοποίησης παράνομων εσόδων και ειδικά όταν πρόκειται για ακίνητα, τράπεζες, μητρώα, κτηματολογίου και το καθεξής. Δεν πρέπει εκεί να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Καλώς. Ε, να ακούμε όμως μία-μία τις ερωτήσεις. Τρεις είναι και οι τρεις θέλουν ερώτηση. Για να δούμε να απαντήσετε στην πρώτη. Απάντηση. Θα συμφωνήσω βέβαια. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια κεντρική δομή του, τελικού, του Μητρώου Τελικών Δικαιούχων, γιατί έτσι όπως έχει σχεδιαστεί τώρα δεν θα έχετε πρόσβαση. Και αν δεν υπάρχει πρόσβαση, μάλλον θα είναι άχρηστο το Μητρώο. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι, εάν οι χώρες, οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι ένα μητρό είναι διαφανές, δεν θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί μόνο όταν ξέρει κανείς ότι μπορεί να κρυφτεί, πηγαίνει σε αυτές τις λύσεις. Η διαφάνεια νομίζω είναι αυτή που θα περιορίσει τέτοιου είδου δραστηριότητε. Για όλα τα άλλα θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε. Ο... Ε, κύριο Σίμαν. Ιβάν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Αυτό που με παρακίνησε να ζητήσω το λόγο είναι η παραπομπή στις ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ότι είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην νομοποίηση από ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Εγώ κατάγομαι από τη Ρουμανία, ε, μάλλον γνωρίζω καλύτερα τι συμβαίνει εκεί. Στη Ρουμανία λοιπόν, μια νεαρά δημοκρατία με νεαρούς θεσμούς και διαδικασίες ακόμη εκμάθησης του πώς μπορούν να σχεδιαστούν σωστά τα πράγματα. Γιατί είχαμε πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε με καινούριο τρόπο μετά την Επανάσταση. Είδαμε πολλές χρηματοοικονομικές ε, μεταφορές, εμβάσματα από την ε, Ρουμανία προς άλλες χώρες και νομίζω ότι πάνε από τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τις μεγάλες επιχειρήσεις των δυτικών κρατών. Το σύστημα με την ε, μεταφορά, το, price, το, το transfer pricing, την κατά μεταφορά τιμολόγηση, την ενδομιλική τιμολόγηση, για να πάνε τα χρήματα αυτά στο Λουξεμβούργο, στην Ιρλανδία, τέλο πάντων σε άλλε χώρε. Και ταυτόχρονα είδαμε και μεγάλου όγκου μέτρητών να μετακινούνται μέσω της Τουρκίας Είδαμε πολλούς από τους πιο διθαρμένους τη Ρουμανία να έχουν μεγάλες επενδύσεις στο Ντουμπάι και άλλες ε, υπεράκτιες άλλου υπεράκτους προορισμού. Συμφωνώ μέσα ότι ενιαία λύση για κάθε περίπτωση, για όλε τι περιπτώσει δεν υπάρχει. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν χώρε δυτικέ οι οποίε εποφελούνται από την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. γιατί χρήματα παράνομα αποκτηθέντα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης νομιμοποιούνται και βγαίνουν πιο καθαρά και πιο ασφαλή σε πιο καθαρές και ασφαλείς και ανεπτυγμένες οικονομίες εμφανίζονται ως ε, καλές επενδύσεις και κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. Άρα νομίζω δεν πρέπει τόσο να, να δεχόμαστε ότι όλοι αγωνίζονται κατά τις νομοποίησεις γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες εποφελούνται. Άρα, ερωτώ, τα, τα κράτη-μέλη πόσο είναι αποφασισμένα να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη νομοποίηση παράνομων εισόδων, γιατί εγώ δεν βλέπω τέτοια βούληση αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, Όντως, ε, η, η, μία από τους διδακτορικούς μας φοιτητές, η Ανδριάννα Ηλιάνου, ήταν ε, Ρουμανά και επομένως ήξερε πολύ καλά την κατάσταση στη Ρουμανία. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια απο τους διδακτορικους μας φοιτητε η ανδριαννα ηλιανου ηταν ρουμανα και επομενως ηξερε εμβασμάτων, που άρα χρησιμοποιεί πολύ το έμβασμα για την ε, νομοποίηση, ε, ενδομιλικές συναλλαγές, όντως, και χωρίς να επενήσουμε ότι η Ρουμανία δεν προβαίνει σε νομοποίηση, έχει χαμηλότερους όγκους, γιατί Αλλιώς, ε, άλλα είναι τα ποσά που μπορεί να μεταφέρει μέσω εμβασμάτων και αλλιώς ε, τα ποσά που μπορεί να είναι μέχρι και 3 εκατομμύρια μπορεί μέσα μια μέρα να διακινηθούν. Και αυτό εννοούσα όταν είπα ότι πρέπει και τα χρηματοπιστωτικά κέντρα αυτά να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχει και αυτό που αναφέρατε εσείς. Είναι εμφανής η υποκρισία των κρατών που ε, προβαίνουν στη μεγαλύτερη, στους μεγαλύτερους όκους νομοποίησης, ενώ είναι και αυτά που εποφελούνται περισσότερο από την νομοποίηση και ταυτόχρονα την καταγγέλουν. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια κοινή συμφωνία, ότι είναι τεράστια η ζημιά που κάνει η νομοποίηση για όλους. Αυτό ακόμα δεν έχει περάσει σε μήνυμα. Μην, μην νομίζει κανείς ότι είναι ένα ε, έγκλημα χωρίς θύμα. Είμαστε όλοι θύματα αυτού του εγκλήματος και πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει στη διαμόρφωση ομόφωνης θέσης και ιδεών. Οι χώρες αυτές που το περισσότερο, συμφωνώ, ότι θα πρέπει να στηρίζουν και να επιδοτούν τις χώρες που υποφέρουν. Γιατί να καταπολεμήσουν δηλαδή οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης την νομοποίηση ενώ η Δυτική Ευρώπη υποφελείται από αυτήν. Πρέπει να εξεταστεί και η λύση κάποιων μεταφορών κονδυλίων προς τις ανατολικές χώρες για να τις στηρίξει για να είναι προς όφελος όλων ο αγώνας αυτός για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης. Αλλά όπως είπατε, τη Ρουμανία την έχουμε ως ιδιαίτερο στόχο μελέτης, την έχουμε ε, εκτεταμένα μελετήσει. Έχουμε πάει και για τις διακοπές μας εκεί για να τη δούμε από κοντά. Ο κύριος Δεμάση. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Και χαίρομαι που ε, ενέπνευσε και τόσα διδακτορικά για τις υπεράκτιες. Δύο πτυχές με εντυπωσιάζουν πρώτα απ' όλα. Γνωστό το φαινόμενο βεβαίως. Η αδιαφάνεια των, της οποίας χαίρουν οι υπεράκτιες και εξακολουθούν να χαίρουν μας κρύβει και τα ποσά και τους όγκους αυτό είναι και η δυσκολία, αυτή είναι και η δυσκολία που έχουμε στην ε, λήψη αποφάσεων πολιτικών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο αξιόπιστα στοιχεία. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ότι η Ευρώπη είναι η ίδια ε, εμπλεγμένη σε όλη αυτή την υπόθεση και δεν μπορεί να κατηγορεί μόνο τον Παναμά ή κάποιε άλλες υπεράκτιες. Οι περιπτώσεις που αναφέρατε επίσης με υποθέσεις που εκδικάστηκαν στις κάτω ε, από εμπόριο ναρκωτικών και που περνούν μέσα από τράπεζες, δεν γίνονται δηλαδή μέσα από μικροπληρωμές, πολλές φορές φτάνουν μέχρι και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πρέπει να το κοιτάξουμε το δίκτυο αυτό, διότι έχουμε κάποιες ενδείξεις από τράπεζες ότι υπάρχει και απευθείας χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Εγώ είμαι Γερμανοϊταλός βουλευτής και έτσι έχω τα πόδια μου σε δύο βάρκες. Τη μία που έχει την ε, καλύτερη επάνδρωση για την καταπολέμηση της ομοποίησης στην Ιταλία και την άλλη που έχει λιγότερη, την λιγότερη επάνδρωση στη Γερμανία. Από την άλλη η Γερμανία μας λέει ότι, αν είχε, ότι έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις, έστω και με ε, χαμηλό αριθμό υπαλλήλων ε, στις υπηρεσίες καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και άρα δεν θα χρειάζονταν περισσότερους. Αλλά εάν ένα ε, αδίκημα έχει διαπραχθεί σε μια δικαιοδοσία άλλη, σε ένα ξενοκράτος. Ε, είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε την πορεία του χρήματος αν δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Και δείξατε στη διαφάνειά σας ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση στη Γερμανία εντωμεταξύ. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα καλά ποια είναι η εικόνα γιατί διαπιστώνω ότι από προσωπική εμπειρία ότι όταν πρόκειται για αδικήματα που έχουν διαπραχθεί σε ξένες δικαιοδοσίες, σε ξένα κράτη, δεν έχουν τέτοια ε, βία να παρακολουθήσουν τις υποθέσεις αυτές οι Γερμανία. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Για δε το θέμα αυτό το οποίο άλλωστε Μα απασχολεί και με την αναθεώρηση της οδηγία. αν θα πρέπει το βασικό έγκλημα του του κατοφένς να ε, συμπεριληφθεί. Προβάλλεται μερικές φορές ε, το επιχείρημα ότι να μπορεί μια νοικοκυρά σε μια χώρα στην, ε, στη Γερμανία να ξεχάσει να, να καταθέσει την ε, ε, φορολογική της δήλωση και να βρεθεί στα, πίσω από τα σύνδεδρα μιας ε, σουηδικής φυλακής. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το παράδειγμα που μας ενδιαφέρει. Δεν μιλούμε για τέτοιε περιπτώσεις. Πρέπει όμως να εντοπίζεται ο τελικός δικαιούχο και κάτοχος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταγράφεται μεν, αλλά εάν πάντοτε δεν είναι δυνατό αυτόν, λένε κάποιοι, θα πρέπει να ορίζεται ο διαχειριστής και το όριο που ορίζουν σχετικά υψηλό για μένα. Εγώ θα έλεγα μπορεί να υπάρχει ένα όριο χαμηλότερο όμως, αλλά ή μη τι άλλο θα έπρεπε να καταγράφονται οι 10 επιφανέστεροι ή πιο σημαντικοί κάτοχοι. Τι θα λέγατε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα. Ήταν ε, ε, η αστυνομία η ε, αστυνομική FIU, η αστυνομική μονάδα οικονομικών μυστικών πληροφοριών. Όταν η Γερμανία έχει 20.000 ε, ε, αναφορές παράνομων συναλλαγών πρέπει να τις διαρευνήσει όλες. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά με την Ολλανδία όπου έχουν τη δυνατότητα επιλογής στη Γερμανία ο μικρός αριθμός ε, αναφορών έχει να κάνει με το κατά πόσο δηλώνεται κάτι στην αστυνομία ε, γιατί εκεί είναι μια πολύ σοβαρή πράξη, δεν είναι απλώς μια καταχώρηση σε ένα φάκελο. Γι' αυτό η Γερμανία ε, κρίθηκαν ότι δεν υποβάλλουν αρκετές αναφορές. Στη συνέχεια, τους είπαν, ε, συνέχεια είχαν περισσότερες αναφορές. Αλλά μετά είπαν ότι αυξήθηκε ο αριθμός του ξεπλήματος. Ε, άρα υπήρχαν πάλι κάποια σφάλματα. Ε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γερμανία προσπαθεί να απαλλαγεί αυτό, αυτό το υπερβελικά αυστηρό νομικό σύστημα που, στο οποίο ασφικτιά. Για τους Γερμανούς η, η, η ανταλλαγή πληροφορών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εάν ε, έχουμε διεθνή συνεργασία, γιατί δεν ήθελα να έχουν διεθνή συνεργασία, γιατί στην περίπτωση αυτή, εάν ε, αναγνώριζαν, εντόπισαν κάποιον ε, ξένο ε, αλλοδαπό, θα είχαν ακόμα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Εγώ προσωπικά ε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να οριστεί ένα κατ κατόφλιο ε, ε, ας πούμε 100.000 ευρώ ε, ούτως ώστε να οριστεί πάνω από αυτό το κατόφλι παράνομη πράξη. Δηλαδή να θεωρηθεί απαράδεκτο κανείς να μην δηλώνει ας πούμε τις 100.000 ευρώ ως κατόφλι ενδεχομένως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, ίσως το κατόφλι αυτό θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό αλλά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για ένα τέτοιο όριο πέραν του οποίου ε, η πράξη αυτή θεωρεί, μπορεί να θεωρηθεί κακούργημα ή σοβαρή αξιόπινη πράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Εξετάζοντας την αξιολόγηση της οδηγίας, λέτε ότι δεν υπήρξε πολιτική συνδρομή από ορισμένες χώρες. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση, Ποιος είναι υπεύθυνο όταν υπάρχουν τέτοιου δυσκολίες. Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη. Είναι πολιτική ευθύνη, είναι διοικητική ευθύνη. Ε, πού ακριβώς εντοπίζονται τα ελλείμματα τα οποία αναφέρατε. Γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει πολιτική αντίσταση εκ μέρου των ο, χωρών. Οι κυβερνήσεις ενισχύουν, είναι υπέρ αυτής της εργασίας. πού εντοπίζονται ακριβώς τα ελλείμματα στην εφαρμογή και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτά. Δεύτερον, έγινε λόγος για διαφάνεια, για πρόσβαση στα μητρώα κλπ, στην ε, ανταλλαγή πληροφοριών και κλπ. Αλλά ε, γνωρίζουμε ότι ήταν εδώ στην Επιτροπή μας και μας είπαν ότι και αυτοί προσπαθούν να εκπονήσουν κάποια συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Βέβαια, αυτό είναι ένα πολιτικό οργανισμό, ο οποίο πρέπει να κάνει κάποιες συμβιβασμού. Κατά την δική αξιολόγηση, ποιο θα ήταν ο πιο αποτελεσματικό τρόπο να γίνεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, ε, ε, τι μπορεί να γίνει στο επίπεδο του ΣΑΠ, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ήδη. Καταρχήν, η πολιτική αντίσταση αφορούσε μόνο την τρίτη οδηγία γιατί ήδη είχαν εφαρμοστεί αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική αντίσταση ε, στην νομοποίηση παράνομων εσόδων. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ε, η αντίσταση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε, στην βραδύτητα με την οποία οι τράπεζες ε, παρέχουν στοιχεία και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν κυρώσεις από την FATF. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει ε, ξεκάθαρο στις ε, κυβερνήσεις ότι με τον τρόπο αυτό διαβρώνεται το πολιτικό μας ε, και οικονομικό σύστημα και νομίζω ότι τα έγγραφα του Παναμά βοήθησαν στην περίπτωση αυτή γιατί κατέδειξαν πόσο διεφθαρμένες είναι πλέον οι πολιτικές ελίτ, οι οικονομικές οι ελίτ ορισμένων χωρών. Τώρα, ποιος θα πρέπει να αναπτύξει αυτά τα εργαλεία για τη διαφάνεια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ήδη να αναπτύξει τα δικά της ε, εργαλεία ανταλλαγή πληροφοριών, ούτω ώστε να είμαστε ισότιμοι εταίροι με τον ΩΣΑ. Αλλιώς ε, ενδεχομένω έχουμε κάτι το οποίο να μην ε, ταιριάζει στις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Χάγη ε, υπάρχει ένα πολύ καλό τεχνικό δέκτυο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ε, εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την Άννα Γκόμες και μετά θα πάρουμε μία ή δύο ερωτήσεις και θα πρέπει να ολοκληρώνουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Χθες ακούσαμε στην κυρία Μπρουκ Χάρεκτον, η οποία είπε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση μπόρεσε να ε, ενισχύσει τη συμμόρφωση εκ μέρους των τραπεζών. Ε, ε, εσείς από τη δική σας μεριά τι κάνατε σε σχέση με αυτό. Όταν συζητούμε την οδηγία υπάρχει αυτός ο κατάλογος των ε, ΠΕΠΣ, των πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων. Αλλά πολύ συχνά είναι εξαιρετικά ανακριβής αυτός ο κατάλογος. Η Επιτροπή Ε, είπε ότι θα, πρέπει, θα έπρεπε οι χώρες μέλη να καταρτήσουν τους δικούς τους καταλόγους με αυτά τα άτομα. Ε, και είπε ότι είναι εφικτό. Αλλά ορισμένες χώρες ε, πρόβαλαν άλλα επιχειρήματα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, την, να ενισχύσει τη συμμόρφωση τουλάχιστον όσον αφορά τα πέπτα άτομα αυτά. Όσον αφορά τη δεύτερη απάντηση για το ΠΕΠΣ, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όντως θα βοηθούσε Τώρα κατά πόσο είναι δυνατόν, εγώ νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες χώρες ε, να το κάνουν. Δηλαδή μπορεί κανείς να συμμετάσχει ή όχι, αλλά τουλάχιστον να αρχίσουν ε, οι χώρες να κάνουν το πρώτο βήμα ε, και οι χώρες οι οποίες θέλουν να έχουν αυτόν τον κατάλογο να το ξεκινήσουν. Το δεύτερο είναι ότι είμαι υπέρ ενός ε, white list ε, και ένας λόγος είναι γιατί νομίζω ότι αρκετά με την τιμωρητική ε, διάθεση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε την συμμόρφωση και νομίζω ότι οι περισσότεροι χώρες, ο κόσμος αντιδρούν καλύτερα στα θετικά στοιχεία και όχι στα αρνητικά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι καλύτερα να αναφέρονται τα, οι επιτυχίες όσον αφορά την καταπολέμηση του, της νομιμοποίησης ε, ε, και αυτό νομίζω ότι θα ε, δώσει έτσι μια γενικότερη θετική ατμόσφαιρα και θα ενθαρρύνει τον κόσμο. Ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα πάρα πολλά άσχημα στοιχεία για τα πάντα. Επομένως, εάν μπορέσουμε θετικά πρόσημα να βάλουμε μπροστά από αυτές τις διαδικασίες θα είναι πολύ καλό. Ε, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν ε, ερωτήσεις, η Κομισιόν, ε, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση για την τυπολογία των FIUs, αυτών των μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Επίσης υπάρχουν ε, καλές ε, πρακτικές, βέλτιστες ε, πρακτικές, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποιες υβριδικές τεχνικές δεύτερον και σε σχέση με αυτό που είπατε για πιο θετική προσέγγιση. Πριν από δύο μέρες είχαμε μια ακρόαση στην Επιτροπή ΠΑΝΑ και ε, έγινε αναφορά ότι ε, δεν υπάρχει έτσι μία, ε, μία από την πλευρά των εμπλεκομένων πολύ θετική διάθεση έτσι ώστε να καταπολεμήσουν πραγματικά το ξέπλυμα. Έχετε κάποια στοιχεία να δώσετε. Εδώ βρίσκομαι, στα αριστερά σας. Ε, ε, είδαμε ένα στοιχείο της ε, μελέτης του επιδιδακτορικού φοιτητού και σύμφωνα με τα νούμερα έκανα τη διαίρεση και φαίνεται ότι η κάθε συναλλαγή αναφέρεται στα 15 εκατομμύρια γιατί μου φαίνεται λίγο πολύ. Τελευταία ερώτηση. Καλησπέρα σας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα παραπάνω όσον αφορά την Δανία. Ε, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς μπορεί κανείς να ασκήσει δίωξη εναντίον κάποιου για ξέπλυμα χρήματος εάν δεν έχει αποδειχθεί ότι το χρήμα ήταν ευρώμικο. What Όσον αφορά την θετική συμμόρφωση ή συμμόρφωση μέσω θετικών ε, παραδειγμάτων, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σύστημα ε, ορθής ε, αναφοράς, reporting, ε, αυτή είναι η έννοια ε, της ε, λευκής, του λευκού αρχείου ή του λευκού μητρώου white list μία λίστα καλών πρακτικών, βελτίστων, αντιμετωπίσεων, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα, τα κατάλληλα. Έχετε δίκιο. 15 εκατομμύρια αλλά είναι αλήθεια ότι ε, στις ε, κάτω χώρες υπάρχουν μερικές συναλλαγές ε, οι οποίες αφορούν πολύ μεγάλες εταιρείες αλλά μπορώ να τον ρωτήσω εάν πραγματικά αυτά τα 15 εκατομμύρια αναφέρονται σε κάθε μία μεμονωμένη συναλλαγή ίσως εννοούσε το σύνολο και από στατιστικά βγαίνει αυτό το πηλίκιο το πηλίκον. Πάντως να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ε, δουλεύει με πάρα πολύ ε, σωστό τρόπο. Λοιπόν, για τη Δανία θα πρέπει, αυτό, θα πρέπει το ίδιο το άτομο, ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο ελεγχόμενος να αποδείξει ότι είναι ε, καθαρά τα χρήματα. Δεν έχει ε, η εισαγγελία την υποχρέωση να δείξει ότι είναι βρώμικα τα χρήματα. Υπάρχει αυτή η αντιστροφή, όπως σας είπα, του βάρους της απόδειξης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αγαπητή κυρία Χούγκερ, για την παρουσία σας και τα τόσα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μας είπατε και τα οποία αποτελούν τροφή για σκέψη. Ελπίζω ότι θα διατηρήσουμε επαφή. Ε, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε.